ευχαριστούμε ως Συμβούλιο με, το, με την Κομισιόν αλλά και με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Και... εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αγγέρη, έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος κατόπιν αυτής της συζήτησης που θα ψηφίσουν αύριο το μεσημέρι. Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου και η πάντηση εκπροσώπου Ένωσης Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας και η ε, Αντιπροέδρου της ε, Επιτροπής όπως είπαμε για την κατάσταση στη Συρία, Μπαχρίνη και η Εμένη. Όμως ε, ε, από πλευράς της θα μιλήσει τώρα ο Υπουργό Εξωτερικών της Προεδρεύουσας χώρας της Ουγγαρίας, ο κύριος Νέμεθ. Μόλις καθίστε με την ησυχία σας και θέτη μας να μας μιλήσετε. speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. Ναι, από εκεί μιλήστε πάνε καλά. Α, παρεξήγησα. Δεν κατάλαβα Πώς τα πού πηγαίνατε. Mr. Bennett, try Yo, yo, yo. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Νέμεθ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ήρθα σήμερα για να σας παρουσιάσω τις ε, παρατηρήσεις μας, τα σχόλιά μας ε, και εκ μέρους της ε, Κάθριν Άστον, της ε, προσώπου για το τι γίνεται εις Σύρια, εις Μπαχρέν και εις Ιεμένη. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν εξελιχθεί ε, σε κάποιο κρίσιμη κατεύθυνση διότι η κατάσταση επιδεινώθηκε στη Συρία και η, κατάσταση που είναι επίσης όσο πάει και βαραίνει παρά το ότι η αιματοχυσία κάπως έχει συγκρατηθεί. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί αυτά τα οποία γίνονται στην ευρύτερη περιφέρεια με μεγάλη προσοχή και αυτό άλλωστε επαληθεύεται από μία σειρά ε, συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Έχουμε επίση τι επίσημε δηλώσει αλλά και τα συμβόλαια του Συμβουλίου. Πέραν όμω όλων αυτών, η Βαρόνη ε, μονίμω έχει επαφή με κάποιου ε, πάρα πολύ σημαντικού παράγοντε και ε, συντελεστές του παιχνιδιού στην περιοχή αλλά και εκπροσώπους αυτών των χωρών και αυτό γίνεται άμεσα με τηλέφωνο με εκπροσώπους μας στις χώρες ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όποτε αυτό είναι δυνατό και όπου είναι δυνατόν αυτό να βοηθήσει πάντως η κατάσταση σε κάθε χώρα είναι διαφορετική και επομένως απαιτείται μια αντίδρασή μας που να είναι στρατηγική να έχει προηγηθεί όριμη σκέψη και θα πρέπει επομένω να δηλάβουμε υπόψη ότι τα γεγονότα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και άρα θα πρέπει να ενεργήσουμε επί τη βάση κάποιων βασικών αρχών και να σα αναφέρω ε, τρεις τέτοιε αρχες αρχές. Πρώτα-πρώτα καταδικάζουμε και απορρίπτουμε την βία. Οι μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες θα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό στα δικαιώματα τη ελευθερία και με ειρηνικό τρόπο. Δεύτερον, θέλουμε να προωθήσουμε το διάλογο, διότι οι πικρίε, οι διαφορέ θα πρέπει πάντοτε με ειρηνικό και υπεκοδομικό τρόπο να αντιμετωπίζονται και θα πρέπει αυτοί που πρέπει να είναι έτοιμοι να καθίσουν στο τραπέζι και να αφήσουν στην, στην άκρη απαγορευτικέ ε, προκαταλήψει. Και τρίτον, ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει όσον αφορά τι ε, οικονομικέ μεταρρυθμίσει και τι πολιτικέ να έρχονται από τα μέσα από κάθε χώρα. Ξεκαθάρισε η Ένωση ότι προτίθεται να υποστηρίξει ε, όποτε τη ζητηθεί ε, αυτές τις κινήσεις. Τώρα θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να μιλήσω για αυτές τις ε, τρεις χώρες για τις οποίες συζητούμε. Πρώτον, Μπαχρέιν. Παρά το ότι οι ομαλότης, ε, οι φυσιολογικοί ρυθμοί της ζωής ξαναγύρισαν, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ κρίσιμη. Συνεχίζονται οι συλλήψεις, διάφορα φυσικά πρόσωπα συλλαμβάνονται, ε, παρά το ότι το μόνο που κάνανε ήταν να ασκήσουν το δικαίωμα τη ελευθερία έκφραση. Όπως και γίνεται και αλλού στην περιοχή, η Ένωση και η ίδια η ψηπάτη εκπρόσωπο, κατεδίκασαν ε, κατηγορηματικά την βία στον Μπαχρέιν και απίθαναν έκκληση στις αρχέ και όλους του εμπλεκόμενου να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μοίρα τη ελευθερία, όπως επίσης και τη διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα. Επίσης, επανειλημμένα έχουμε καλέσει τις ε, αρχές της χώρας αλλά και την αντιπολίτευση να καθίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο και η Πάτη Πρόσωπος επίσης ήρθε σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς για αυτό το λόγο. Ε, χωρίς να γίνουν συγκεκριμένα διαβήματα ούτως ώστε να μιλήσουν τα αντίπαλα μέρη ε, χωρίς προκαταλήψεις ε, με καλή θέληση να μιλήσουν τότε ε, οι πιο ριζοσπάστες τα πιο ακραία στοιχεία θα κυριαρχήσουν θεωρούμε επομένως ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την περιφερειακή σταθερότητα και ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε αυτή την σταθερότητα να την διαφυλάξουμε είναι ο διάλογος. Αυτό είναι το μήνυμα της υπάρξης εκπροσώπου και αυτό θα κάνει όταν έρθει η ώρα να συναντήσω τους υπουργού ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου το οποίο θα γίνει πάρα πολύ σύντομα αυτόν τον μήνα. Ε, στην Συρία τώρα ε, οι διαδηλώσεις, οι λαϊκές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας λαμβάνουν χώρα σε πάρα πολλές πόλεις από τα μέσα του Μαρτίου και η καταστολή ήταν βία, αλλά θεωρήθηκε απαράδεκτη. Η Πατήκρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει πάρα πολλά διαβήματα προς τις αρχές της χώρας, ώστε να σταματήσει αυτή η βία να σεβαστούν το δικαίωμα του λαού εις ε, διαμαρτυρία και να αφουγκραστούν τα, τα, τα νο, θεμητά τους αιτήματα. Ο λαός της Συρίας ε, αξίζει αυτές τις προσδοκόμενες ε, πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συναθρίζεστε, την ίδρυση κομμάτων, την, την συμμετοχή στο Υπουργό αλλά και στην διακυβέρνηση της χώρας. Άλλωστε η ομιλία του Πρόεδρου Ασάντ ε, προς ε, τη χώρα στις 30 Μαρτίου είπε ότι ε, οτιδήποτε άλλο εκτός από το να πει συγκεκριμένο προδιάγραμμα για τέτοιες μεταρρυθμίσεις και υλοποίηση των όσων έχουν εξαγγελθεί. Επομένω, η Ευρωκοινή θα συνεχίσει να πείζει τη χώρα ούτω ώστε η Συρία να προβεί αμελητή σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Μα τι, ένα τηλέφωνο κάπου χτυπάει μέσα στην αίθουσα. Great. All right. Θα συνεχίζουμε επομένω να πιέζουμε τη Συρία ούτω ώστε να υλοποιήσει αυτέ τι μεταρρυθμίσει για αυτό να γίνει αμελητή. Ε, Επίση θέλουμε να είναι ουσιαστικέ, πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ. Να μην είναι εμβαλωματικέ, να μην είναι ε, ε, σαν πρόφαση να είναι, ε, οι προσχηματιές να είναι σοβαρές και επίσης να εφαρμοστούν τόσο και εμείς θα παρακολουθήσουμε ό,τι κάνει η κυβέρνηση από κοντά. Θεωρούμε ότι η συγκρότηση της νομικής επιτροπής θα οδηγήσει εις θέσπιση νέας νομοθεσίας, ούτως ώστε να αρθεί η κατάσταση πολιορκίας και να υπάρξουν εγγύσει για ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συνεχίσει να πιέζει την ηγεσία τη χώρα. Δημοσίω και ατύπω, ούτω ώστε να σταματήσει η άσκηση βία καταστολή κατά των ε, διαδηλωτών. Επίση, είναι σημαντικό ε, να περάσουν από δίκη αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ε, βία, για τα θύματα που έχουν σημειωθεί αλλά επίσης θα πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και κυρίως οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμένη. Η κατάσταση προβληματίζει πάρα πολύ. Η είπατε εκπρόσωπος ε, προέβησε κάποιες ανακοινώσεις κατόπιν τη καταδίκη αυτών των βίων γεγονότων του 18 Μαρτίου. Ήταν ξεκάθαρα αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση για του στόματό τη και είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών τη 21η Τρίτου. Επαναλαμβάναμε γιατί καταδικάζουμε την άσκηση βία και καταστολή. Επίση, η τριτου Επαναλαμβάνομαι γιατι καταδικαζουμε Ένωση τοποθετήθηκε ε, υπέρ ε, της ε, απονομής δικαιοσύνης και της, του καταλογισμού των ευθυνών σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες. Πάντως δεν είναι σαφή η στάση των αρχών της χώρας. Γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή, ήρθε σε επαφή η πρόσωπος με τον πρόεδρο Σαλέξ στις 33 και είπε ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σταματήσει την περαιτέρω αιματοχυσία και είπε ότι η άποψή της είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο είναι να υπάρχει κάποιο είδους μετασχηματισμός αξιόπιστος και γρήγορος και να ξεκινήσει αυτή η δικασία επίσης αμελητή η δε συνταγματική μεταρρύθμιση θα πρέπει να έχει ως αφετηρία κάποιες δεσμεύσεις συνεπείς, ουσιαστικές και οι οποίες δεσμεύσεις να υλοποιηθούν ο χρόνος πιέζει και τελικά τα θύματα της κατάστασης είναι ο λαός της χώρας και για αυτό ε, συνεργασία με άλλους ε, παράγοντες της διεθνούς σκηνής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εμπλέκεται και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κρίση στην Ιεμένη ε, και να πασχίσει να βρεθεί μια διέξοδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την προσοχή σας και περιμένω πώς και πώς παρατηρήσεις σας αλλά και ερωτήσεις σας. Ο πρόεδρος ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Και τώρα ε, Ποιο το ήταν ο Μπρο Μπρόκ, ο Σαλαφράγκα. Κύριε Σαλαφράγκα, συγχαρητήρια και στου δύο. Α, στον κύριο, στον κύριο ε, Μπρόκ, γιατί βλέπω συγχαρητήρια για την μεγάλη νίκη τη ομάδα σα τη ΣΑΛ και βλέπω φοράτε και το κασκόλ. Και βέβαια αυτό το πετύχατε με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον Ισπανό Ραούλ. Και τώρα όμω, ο κύριο Σαλαφράγκα θα λάβει το λόγο για ένα λεπτό και μισό για του Ευρωπαϊκού Λεγόμενου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ για όλα όσα είπατε όσον αφορά την ομάδα του κύριου Μπρόκ. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ε, τα όσα μας ενημερώνει η πατηκπρόσωπος για την εξέλιξη των γεγονότων σε αυτές τις χώρες. Και νομίζω ότι οφείλουμε να γνωρίσουμε τις καταπληκτικές προσπάθειες που έγιναν ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να προωθήσουμε σε αυτές τις τρεις χώρες ε, τις δημοκρατικές αρχές. Αύριο δεν πρόκειται να εγκρίνουμε το σχετικό κείμενο και όλες οι πολιτικές ομάδες θα το επιψηφίσουν. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να θέσω κάποια ερωτήματα. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, διαβάστε αυτά τα ερωτήματα στην υπάτη εκπρόσωπο. Πρώτον, διάφοροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός πισωγυρίσματος όσον αφορά τις εξελίξεις για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική, εξωτερική και ασφάλειας. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στην πολιτική συνεργασία. Άρα δεν ωφέλησε η συνθήκη τη Λισαβόνα. Έχουμε εδώ πέρα μπροστά μα μια αντίφαση. Δηλαδή, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι παρουσία τη Ένωση σε αυτέ τι Θα πρέπει όμω επίση να κάτσουμε και να σκεφτούμε ο μετασχηματισμό που θα γίνει, πού θα οδηγήσει. Πάντω εμεί θα πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντε. Καλά. Τα είπε η κυρία Στον. More for more. Άρα, να κάτσουμε και να σκεφτούμε αν τα κράτη-μέλη προτίθενται να αυξήσουν την πρικοδότηση για αυτά τα διαδήματα, για αυτέ τι κινήσει μα, για την παρουσία μα σε αυτές τι χώρε. εμεί ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και τώρα. για Σοσιαλιστική Ομάδα για δύο λεπτά έχει τον λόγο η κυρία Βερονίκ Ντε Κάιζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <coughs> Έχουμε συνείδηση των ε, εντατικών ε, διπλωματικών προστατευτικών της κυρίας ε, Άστον. Ξέρουμε ότι συνεχίζει και επίση έχουμε συνείδηση και των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στη Συρία, την Ιεμένη, τον Μπαχρέιν. Δεν υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίε ε, με ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φερρυπίνη. Έχουμε δηλαδή πολύ περιορισμένο ε, πεδίο πίεση. Αλλά θα ήθελα να πω τα εξή. Πρώτον, σε σχέση με τις ε, προσδοκίες των λαών, των ανθρώπων που κατεβαίνουν στους δρόμους, και αντιμετωπίσουν τι επιθέσει των ελεύθερων σκοπευτών. Πρέπει σε αυτού του ανθρώπου να συμπαρασταθούμε και να ζητήσουμε πάση θυσία το πέρας των ανθρωπραξιών. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι και το είδα και σήμερα με τους Σύριους είναι ότι προσπαθούν να θέσουν ένα τέρμα στη βία. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν δεν έχουμε αντίστοιχε συμφωνίε με τη Συρία, θα πρέπει με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μα ω οπλοστάσιο κυρώσεων, εάν είναι απαραίτητο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή τη βία. Δεύτερον, οι χώρε εν γέννη, ειδικά του Περσικού κόλπου αλλά και η Λιβύη βεβαίω, είναι ακριβώ οι χώρε αυτέ οι οποίε εμεί εξοπλίσαμε. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να ελέγξουμε τους εξοπλισμούς και κυρίως ε, εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να τις μετατρέψουν την αποθήκη εις βάρος των πολιτών. Και τρίτον, προδιαγραφές. Με τον Μπαχρέν ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί, ήμασταν πολύ πιο αυστηρή σε σχέση με άλλες χώρες. Ξέρω ότι το Μπαχρέιν είναι μια πολύ λεπτή κατάσταση. Έχει αποστείλει ε, το Συμβούλιο του Περσικού με τη Σαουδική Αραβία στρατεύματα και μας βοηθούν κιόλα το Συμβούλιο του Περσικού και η ε, Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν μπορούμε να σταθμίσουμε τη τιμή του βαρελιού του πετρελαίου με την υποστήριξη προς την, ε, μια κυβέρνηση ενδεχομένω της Λιβύης και το τίμημα της σιωπή ε, για τους ΣΥΙΤΕΣ τους οποίους καταπιέζει και καταδυναστεύει η κυβέρνηση του Μπαχρέν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ εκ μέρους των φιλελευθέρων για δύο λεπτά η κυρία γιατί με Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι οργή. Εχθές στη συνεδρίαση της ομάδας από τρεις μάρτυρες που προερχόταν από τον Παχρέν, τη Συρία και τη Λιβύη μαρτυρίες. Ήταν από την ε, Human Rights Watch, από την ε, Διεθνή Αμνηστία. Ακούσαμε ιστορίες λοιπόν που είχαν δύο αυτοπές μάρτυρες και αισθάνθηκα οργή. Η επιστολή της κυρίας Άστον δεν είναι στρατηγικό κείμενο. Είναι μόνο ένα άλλο πρόγραμμα, ένα επιπλέον πρόγραμμα Δηλαδή σαν να κάνουμε τα ίδια πράγματα με αυτά που είχαμε και, στην, ε, και σε σχέση με την, ε, την Ισία, την Αίγυπτο ή τη Λιβύη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να ε, συνέλθει εκτάκτο στο Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Πρέπει προς τις τρεις χώρες να ζητήσουμε την λογοδοσία των καθιστώτων για τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ε, δεύτερον, θα πρέπει να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόλυτη εξαγωγή την απόλυτη απαγόρευση όλων των εξαγωγών όπλων προ τι τρει αυτέ χώρε Είναι απαράδεκτο χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη να πολλούν όπλα και εξοπλισμού σε αυτά τα καθεστώτα. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι τα πολιτικά καθεστώτα σε αυτέ τι χώρε. χώρες αποτελούν εμπόδιο στην δημοκρατισμό τους και ήρθε πια η ώρα να ε, καταρριφθούν, να φύγουν και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα και να παγώσουμε τα ε, περιουσιακά του στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό κυρία Φλότχο, η οποία μιλεί εκ μέρου των Πρασίνων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή η είδηση πως αρχίζουν οι λαοί να κινούνται και διεκδικούν ελευθερίες, δικαιώματα και αλλαγή πολιτικού καθεστώτος περισσότερες ελευθερίες. Αυτό αποτελεί και το επίκεντρο των πολιτικών και των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού οράματος και εγχείρηματος. Δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε ενθουσιασμό και να προσφέρουμε την υποστήριξή μας. Ωστόσο, βλέπουμε δυστυχώς ότι υφίσταται σημαντική, σκληρότατη καταστολή αυτές ε, οι αυτοί οι πολίτες ε, πολλές φορές ακόμη και τη ζωή τους πρέπει να δώσουν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό είναι απαράδεκτο λοιπόν. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες αυτούς, τους λαούς αυτούς και όπως ακριβώς αποστήλαμε στρατιωτικέ δυνάμεις στη Λιβύη πρέπει με άλλους τρόπους να προστατεύσουμε τους ε, πολίτες που διαδηλώνουν σε αυτά τα τρία κράτη. Είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις, οι διακηρύξεις, ε, ε, και οι προσδοκίες που, που εκφράζουν οι πολίτες αυτοί είναι θεμητές αλλά πρέπει πλέον τα λόγια που ακούμε να τα μεταφράσουμε και σε πράξη. Πρέπει να δείξουμε στους προσώπους αυτών των καθεστώτων που χρησιμοποιούν άμετρη βία εις βάρος των πολιτών τους για την καταστολή ότι δεν έχουμε πλέον άλλο περιθώριο ανοχής και θα πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δραστηριότητες με αποστολές, με εκθέσεις ε, με κυρώσει έτσι ώστε αυτή η πολιτική ε, ταγή να αντιληφθούν επιτέλους ότι δεν πρόκειται να μείνει ατιμόρυτη αυτή η καταστολή και επιπλέον πιστεύω ότι θα πρέπει κάθε μέτρο που έχουμε να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το απόλυτο blackout ως προς τον τύπο και την ενημέρωση προς τα έξω. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά. Έχουμε μέσα στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την απαγόρευση δημοσίευση ειδήσεων και πρέπει να το θέσουμε σε δράση. Για δε τις ε, κυρώσεις πιστεύω πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κυνηγάμε τον ε, Σύριο Πρόεδρο για να εξασφαλίσουμε τη συμφωνία επανεισδοκής, ε, την υπογραφή του καλύτερα στη συμφωνία επανεισδοκής που δεν μπορεί βέβαια να υλοποιηθεί παρά μόνο επί όρου ενό πολύ αυστηρού προγράμματο και συνεπού προγράμματο ε, μεταρρυθμίσεων στη χώρα αυτή και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών ε, κρατουμένων αντιφρονούντων και των ε, ειρηνικών διαδηλωτών όπως και στις τρεις αυτές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Καρίμ, ρυθμιστές της Ευρώπης. Η κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ, κάθε εδώ και άκουσα τι εγγυρώσει σα και σα άκουσα προσεκτικά, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι απλέ λέξει, πολλέ φορέ πάρα πολύ συμπαθητικέ, αλλά δυστυχώ ε, κενέ λέξει. Όλα αυτά ε, ήταν ε, παθητική εκδήλωση, δεν ήταν κάτι το, το, το δυναμικό και σας άκουσα και προσπάθησα να σημειώσω αυτά τα οποία μας λέτε σε σχέση με αυτά που είχε εξαγγείλει η Πατικροπρόσωπος ότι θα κάνει. Τίποτα δεν βλέπω εδώ. Θα σημείωνα τι αντιστοιχεί σε υποσχέσει αυτά που γίνονται. Τίποτα δεν σημείωσα, τίποτα δεν είπατε, τίποτα δεν υπάρχει το οποίο να αποτελεί ανάληψη πρωτοβουλία. Γιατί έχουμε τόσο κόσμο στη Μέση Ανατολή που προσβλέπουν στην Ευρώπη, ούτω ώστε να του βοηθήσει να ανακτήσουν τα δικαιώματά του. Και τι έχουν μόνο, καινού λόγου. Είχαμε το αυτό το τελευταίο σχέδιο δράση το οποίο προωθήθηκε και υπήρχε κάτι το οποίο απουσίαζε πάρα πολύ και βοούσαν τα ΜΜΕ ότι ε, έρχεται χρήμα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους ηγέτες αυτών των χωρών που τα παίρνουν από το λαό τους και δεν κάνουμε τίποτα για να τους σταματήσουμε. Ισχύουν αυτά. Και αν ε, ισχύουν όλα αυτά, γιατί τελικά έρχεστε εδώ και μας λέτε όλα αυτά τα, τα, τα κενά λόγια. Παρακαλώ, σεβαστείτε λίγο την κατάσταση. Ευχαριστούμε κύριε Σανάδελφε Λεοπρόεδρος και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ματίας για την Ευρωπαϊκή ε, Νοτική Αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ή στην Ιεμένη, ή στην Συρία, αλλά και στο Μπαχρέιν, κοινό παρονομαστή είναι ότι ο κόσμο θέλει ε, δημοκρατία και ελευθερία. Αλλά και έχουμε αυτό το λουτρό αίματο, αυτή την εκτεταμένη καταστολή. Επομένω, θα πρέπει να είμαι θα σαφή, ξεκάθαρη και οπότε, πρώτα-πρώτα, παρακαλώ σταματήστε να πουλάτε όπλα ει αυτέ τι χώρε. Η Ευρώπη συνεχίζει να πουλάει όπλα. Αυτά τα όπλα σκοτώνουν του αμάχου, του πολίτε. Οπότε παρακαλώ, ασήμεθα στο πλευρό και με το πλευρό του λαού και όχι αυτών των καθεστώτων που είναι αυταρχικά καθεστώτα που είναι δικτατορίες. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι η Ευρώπη έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, Από τη, ε, απ τη μια για τις ε, θεμητές φιλοδοξίες των λαών και άλλο για τις εμπορικές συναλλαγές. Στην Λιβύη οι βόμβες κατήργησαν τον ΟΗΕ. Στη, στον Μπαχρέιν δε είπαμε τι έγινε ε, για τη Σαουδική Αραβία και λοιπά συνεχίζεται εκεί πέρα η αυταρχική κατάσταση οι νέοι άνθρωποι ε, έχουν προτάξει τα γυμνά στήθους ή στο στρατό ή στην αστυνομία και εμείς τι κάνουμε μόνο νότες διπλωματικές επαφές δεν είναι σωστό να υπάρχει στρατιωτική επανέμβαση, αλλά επίση ούτε είναι σωστό ο κόσμο να θεωρεί ότι εμεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμεί ευχαριστούμε. Μπέλτερ. Ευρώπη Ελευθερία και Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Συρία Μπαχρέιν και η Εμένη οποιαδήποτε ριζοσπαστική αλλαγή καθεστώτος θα σήμαινε μεγάλη κρίση και για τις χώρες αυτές αλλά και για τις γειτονικέ τους. Και θα έκαναν τα χέρια τους οι Ιρανοί ηγέτες, την Αχμεντινιτζάντ. Και θα χανόταν αυτή η μεγάλη ευκαιρία μιας αραβικής άνοιξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα μαζί με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν αυστηρούς όρους στα καθεστώτα αυτά για την περαιτέρω στη, στο Βαχρέιν δηλαδή, στο καθεστώς του Βαχρέιν για οποιαδήποτε περαιτέρω υποστήριξη. Ε, χρειάζεται εδώ μια προειδοποίηση και όχι μετά από την κρίση. Ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Τελειώνει αυτός ο γύρος ομιλητών με παρέμβαση ενός λεπτού του κυρίου Μέλτσερ των μη εγγεγραμμένων. Στην Ιεμένη, Παχρέν και Συρία δεν προχωρεί τόσο ειρηνικά αυτή η επανάσταση των γιασεμιών. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να συμμετάσχει η κυβέρνηση στις, η κυβέρνηση συμμετάσχουν και να υπάρξει μεγαλύτερη δημοκρατική συμμετοχή. Εάν βέβαια τέτοιε συμφωνίε είναι δυνατόν να γίνουν αλλά και να τηρηθούν, αυτό είναι τελείω διαφορετική υπόθεση. Ιδίω οι μη τηρηθήσει υποχρώσει ε, περί ε, πολιτικών μεταρρυθμίσεων είναι αυτέ που οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση του ε, κόσμου. Η διπλή στρατηγική από τη μια μεριά βίαιης καταστολή των διαδηλώσεων και από την άλλη μεριά μικρών προτινόμενων μεταρρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει εν τέλει σε κλιμάκωση της καταστάσεως στις τρεις αυτές χώρες. Ιδίω με τις ε, διαρκείς ταραχές στην Συρία ε, ξε, ξεκινά και πάλι η ανησυχία από το γεγονός ότι θα μπορούσε να δοθεί περαιτέρω υποστήριξη από το καθεστώς αυτό σε ριζοσπαστικές οργανώσεις όπως η Εσβολάχ. Πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στους μεμονωμένους αγορητές. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζουμε ότι ο Ραούλ είναι μεγάλος ε, ποδοσφαιριστής. Εν πάση περιπτώσει, έρθουμε στο θέμα που μας απασχολεί τώρα. Στα μέρη αυτά του κόσμου. Και παντού βλέπουμε τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου να έχουν σπάσει την απομόνωση και να έχουν γύρει προσδοκίες εκδημοκρατισμού. Υπάρχει ένας νέος ακτιβισμός, ένας νέος τρόπος διεξαγωγής της πολιτικής που αρχίζει και προσελκύει τους πολίτες και ιδίως τους νέους, γιατί οι νέοι έχουν εντονότερα την συνείδηση των ε, τεκτενωμένων από ότι ε, οι πλέον ηλικιωμένοι. Για παράδειγμα, πρόσφατα έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιεμένη, όπως και το Παχρέιν, εκτός από τη Συρία, οι γνωστές ε, κινητοποιήσεις. Χρειάζεται λοιπόν αντίδραση για να πάψει η χρήση βίας από πλευρά των καθεστώτων. Πρέπει να ενισχυθεί η πορεία των χωρών αυτών προς τη δημοκρατία. Αυτά που γίνονται γύρω από τη Μεσόγειο σίγουρα είναι δύσκολο να κατανοηθούν μηνύματα Πρέπει ωστόσο η Ευρώπη να φανεί αλληλέγγυα με τις παρεμβάσεις της και να βοηθήσει την περιοχή αυτή η οποία βεβαίως πάντοτε είναι και εκτεθειμένη σε μεταναστευτικές ροές. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Χάουιτ. Είτε πρόκειται για τις συντονισμένες επιθέσεις των ελευθερών σκοπευτών στις Σανά η καταστολή των ε, διαδηλωτών στην ε, Συρία στις 17 Μαρτίου η επίθεση στο νοσοκομείο στο Μπαχρέιν όπου είναι υποχρεωμένοι να πάνε εκεί οι τραυματίες διαδηλωτές διότι μόνο εκεί υπάρχει τράπεζα αίματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων οπουδήποτε του κόσμου αυτά ε, διακυβεύονται σήμερα ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, από το Συμβούλιο μάλλον των Υπουργών Εξωτερικών, να ζητήσει ε, μη ατιμορρησία, έρευνε και ανακρίσεις για την ε, διαπίστωση των ενόχων. Όταν, μιλούμε, όταν ακούμε μάλλον τις ε, δυνάμεις του Μπαχρέιν ότι χρησιμοποίησαν ε, υποτίθεται μη ε, θανατηφόρα όπλα από ελάχιστη απόσταση ο, πραγματικά ε, σκότωσαν διαδηλωτές πρέπει να ρωτήσουμε που πάνε και τέλος οι αρχές της ε, ε του κυρίου Φούλε για την πολιτική γειτονία πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να υπάρξει όντως μια συμφωνία συνδέσεως με τη Συρία και να ζητηθεί α, ανεμπόδιστη πρόσβαση ε, των ερευνητών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. 1,5 λεπτά. Ο κύριος Λάμστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, άνοιξη στην Μεσόγειο, αλλά χειμώνας στον Περσικό και στη Συρία. Οι εικόνες που βλέπουμε από την βία είναι φρικαστικές εκατοντάδες νεκροί, η Διεθνή Αμνηστία και οι Ηνωμένα Έθνη έχουν κάνει τους απολογισμούς. Οι απαιτήσει είναι ξεκάθαρες και θα πρέπει τι απαιτήσει αυτέ να τι υιοθετήσει και το Συμβούλιο. Ταχύτατα θέλουμε ε, σύγκριση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Τώρα πρέπει να αναλάβει δράση απέναντι σε αυτές τις μαζικές καταπίεσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε πορεία προς την δημοκρατία, χρειαζόμαστε εμπάργκο στους εξοπλισμούς. Εγώ είδα την ομιλία του Προέδρου της Συρίας. Πρόκειται για μια μεσαιωνικού χαρακτήρα ε, δικτατορία που ωστόσο πληρώνει ευρωπαϊκές ε, εταιρείε διαφημίσεων για να την εμφανίζουν ως δίθεν σύγχρονη. Θα πρέπει να ρωτήσουμε και, αυτές, και αυτούς τους οργανισμούς αν πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο. Η εμένη τώρα. Υπάρχει μέγας κίνδυνος διάσπασης βορρά από νότο. Ένα αποτυχημένο κράτος όπως η ε, Σομαλία. Στον κόλπο του Άντεν έχουμε ήδη την επιχείρηση Αταλάντη. Θα πρέπει να ακούσουμε λίγο περισσότερα πράγματα από αυτά που είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Λάμπστορφ. Ένα λεπτό. Η κυρία Φρίντα Μπρέπολς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω πως με έκπληξη καταγράφω τις τρεις αρχές που ανέφερε ο κύριος υπουργό, δηλαδή απόρριψη κάθε μορφής βίας, προαγωγή του διαλόγου, προσπάθεια επίλυση των διαφορών και ενθάρρυνση πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, κάθε έκκληση για διάλογο είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα και μάλλον αποτελεί και δείγμα αναξιοπιστίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε σαφέστερα σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις και αν δεν είναι διθέσιμα τα καθεστώτα να τις επιβάλλουμε. Ερωτώ επίσης πώς διατηρείται σχέση σε πλευρά του Συμβουλίου με τους διάφορους αυτούς ηγέτες και εάν ακούγονται οι παρατηρήσεις μας. Πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα στις ε, εξαγωγές όπλων. Μόνο στην Ιεμένη πάνω από 100 εκατομμύρια ε, ευρώ πούλησαν 8 κράτη-μέλη μόνο το 2010. Πολύ καλό αυτό ε, προς τις επιδόσεις μας εξαγωγές όπλων. Πώς θα πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε για 1,5 λεπτό. Έχει τώρα το λόγο ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για τον Μπαχρέιν, αυτή τη μικρή χώρα που έχει όμως μια στρατηγική θέση και είναι πολύ χρήσιμη θέση της για τις οποίες τον ε, κόλπο αλλά και για λόγους ενεργειακούς και επίσης εκεί πέρα υπάρχει και αυτό το δηληστήριο ε, που αφορά και τη Σοβική Αραβία, πρόκειται για μια στεγματική δημοκρατία και έχει κάποιο κοινοβούλιο και έχει ανεξάρτητη δημοκρατία και είναι τώρα και άλλε μεταρρυθμίσει ε, επίσης είναι πάρα πολύ σύντες στη χώρα. Οπότε και αυτό έχει να κάνει με τις ε, θεμητές προσδοκίες ε, και τις απαιτήσει για μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια ε, να δούμε τι, ποια είναι η πραγματικότητα γιατί υπάρχουν εξωτερικές πιέσεις έχουμε τα, αυτά τα πρόσφατα γεγονότα όμως υπάρχει ο κίνδυνος αποστεθροποίησης ε, σε μια χώρα, ε, σε μια περιοχή που καλύπτει και τη Σαουδική Αραβία και, και εκεί έχουμε του Ιήτε, ε, γιατί ξέρουμε ότι το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χαμάς υποστήριξε Χεσμολάχ στο Λίβανο και, και επίσης επηρεάζει την εσωτερική πολιτική στο Ιράκ και εκεί έχουμε πολλούς ε, Επίσης, αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον, τον, τον, την περιοχή του κόλπου, τότε είναι δυνατόν με το ειδικό τους βάρος να ανατρέψουν την ισορροπία. Επομένως, χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την αξιολόγηση του τι γίνεται στην Μέση Ανατολή και να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των θεμητών προσδοκιών και για περισσότερη δημοκρατία σε σχέση με αυτές τις ε, εξωτερικές ε, επιρροές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο κύριε Όμιρο Ράιτον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα μιλάμε για πολύ διαφορετικά κράτη, κράτη τα οποία έχουν το καθένα το δικό του πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά. Στην Ιεμένη ε, γνωρίζουμε μια μαζική αντίδραση παρά την καταστολή από την αστυνομία στο Μπαχρέιν. Έχουμε κίνδυνο αποσταθεροποίηση όλη τη περιοχή λόγω συμμετοχή ή εμπλοκή του Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Στη δε Συρία η αντιπολίτευση δεν έχει σχεδόν κανένα περιθώριο χειρισμού και φαίνεται ότι το καθεστώ είναι τεθειμένο να λάβει κάθε παρέτο μέτρο για να καταστήλει τι εξεγέρσει. Δεδομένων λοιπόν αυτών των διαφορετικών συνθήκων, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει διμερεί επαφές κυρίως και αυτό με βάση κάποιες συγκεκριμένε αρχές. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελευθερία της πολιτικής διαδήλωσης, έκφρασης πολιτικής άποψης. Ωστόσο όταν διεξάγονται ε, ειρηνικές ε, διαδηλώσεις θα πρέπει να ε, υφίστανται καταστολή οι πολίτες. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Θα γίνει κάποια διεθνή εξέταση τη υπόθεση παραδείγματι του περιστατικού. Και επιπλέον θα πρέπει να ενισχύσουμε, πιστεύω, το διάλογο μεταξύ τη ε, αντιπολίτευση ε, και τη κυβέρνηση. Γιατί η βία δεν μπορεί να αποτελέσει ποτέ λύση. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Εάν το καθεστώ στη Συρία, τον Μπαχρέν, την Ιεμένη, δεν θέλει να εισακούσει τους πολίτες του ή αν δεν σε θέση να το πράξει θα υπάρξουν συνέπειες ως προς τη σχέση μας μαζί τους. Σε αυτό νομίζω θα πρέπει να κάνουμε σαφείς, ε, να λάβουμε σαφείς θέσεις. Και νομίζω πρέπει να συμβάλλουμε συγκεκριμένα με βοήθεια συγκεκριμένη. Θα ήθελα λοιπόν ο Υπουργό να μα πει ποιε είναι οι προθέσει του συγκεκριμένα στην υπόθεση αυτή. Για δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Συρίας φρονώ ότι θα πρέπει στην ουσία να επιμείνουμε με περισσότερες πιέσεις, με πραγματικέ πιέσεις και να φροντίσουμε ώστε να μην εισπράξει στο προσεχέ ε, διάστημα καμία ενίσχυση οικονομική η Συρία. Το ίδιο θα πρέπει να επιδιώξει και η αντιπροσωπεία μα για το Μαστρέκ, κύριε Πρόεδρε, να προσπαθήσει δηλαδή να πιέσει. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε μου. Μου είπαν οι υπαλλήλοι ότι πιέζει πολύ ο χρόνο. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να προσαρμοστείτε στον χρόνο που έχετε ως αγορητές από τις ομάδες σας. Για ένα λεπτό, η κυρία Αναγκόμεθ παρακαλώ. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί στις δηλώσεις και δράσεις μας όσον αφορά τα μέτρα για τη Συρία, το Μπαχρέν και άλλες χώρες στον αραβικό κόσμο διακυβεύεται κάτι παραπάνω από την αξιοπιστία. Η ίδια η αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων που αποστέλλονται, καθώ επίση και για του άνδρες και γυναίκε που διακινδυνεύουν τις ζωέ του να κατεβούν στου δρόμου και να ζητήσουν δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάσταση στον Παχρέν ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αμφίσιμη ε, στάση. Και εδώ βλέπουμε τι αντιφάσει μια εξωτερική πολιτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά λόγω του πετρελαίου και λόγω των όπλων που διατίθενται όχι μόνο στο Μπαχρέν αλλά και σε άλλες χώρες και την παραβίαση των ρητρών για τέτοιου είδους εξαγωγές απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει η ύπατη εκπρόσωπος να προσαρμοστούν ε, οι κυβερνώντες στο Μπαχρέιν ε, ιδιαίτερα με τις διατάξεις αυτές και να σταματήσουν αμέσως τα μέτρα των blackout των μέσων ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκόμεθα. Για ένα λεπτό επίσης στη συνέχεια ο συνάδελφος Μακμίλαν Σκότ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χθε το βράδυ βοήθησα να διοργανωθεί μια ακρόαση επαϊόντων από την περιοχή αυτή και ακούμε ότι στο Μπαχρέιν οι ε, περιπτώσεις αποβιωσάντων είναι 23, στην Συρία 132, στην Ιεμένη τουλάχιστον 63 που απεβίωσαν. Ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα που θα υιοθετηθεί αύριο υποβάλλει κάποιε προτάσει, αλλά πρέπει να πω ότι του προηγούμενου μήνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα για την Ισία, την Αίγυπτο, την Λιβύη. Και το γραφείο μου συνέκρινε μεταξύ αυτών των ψηφισμάτων και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχεδίων για αλλαγές και δεν μου δίνουν ιδιαίτερο χάρος. Χάνουμε τα λόγια μας εδώ, εκτός αν ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακούει και προσαρμόζεται το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν, σε σχέση με την ιστοσελίδα μου, και πιστεύω ότι η συνθήκη της Σαββόνας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθετες ευθύνες. Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα σοβαρά αυτές οι Ευθύνε από τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή και Συμβούλιο. Με την περίοδο αυτή μαζικών αλλαγών στον αραβικό κόσμο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Σαρλάκη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η Συρία, το Μπαχρέν και η Εμένη είναι ε, καθεστώτα που αμφισβητούνται από τους ίδιους πολίτες τους και βλέπουμε ότι έχουν ε, ανεπιφύλακτη υποστήριξη. Μέχρι σήμερα η δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εκδημοκρατισμό είχε απουσία σθένους ε, και αξιοπιστίας. Αν θέλουμε να πετύχουμε πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε άροντας τα, έροντας τα διπλά μέτρα και σταθμά που ισχύουν και να μπορέσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να πούμε ότι είχαμε προσπαθήσει να πουλάμε σε αυτούς ε, όλο, όλο, όλων των ειδών τα όπλα και τώρα εκφράζουμε την θλίψη μας ε, για τα θύματα, για τα αθώα αυτά θύματα που ε, υπήρξαν λόγω αυτών των δράσεων, αυτών των καθεστώτων. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να καταργήσουμε όλες τις συμβάσεις παροχής όπλων σε αυτές τις χώρες και να ζητήσουμε να θεσπιστεί εμπάργο σε όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής η μείωση του, ε, των στρατιωτικών εξοπλισμών θα είναι ένα, μια πρόσθετη αξία που θα επενδυθεί στην ε, δημοκρατική αλλαγή. Η κυρία Μουνίθα ε, τελευταία που θα παρέμβει ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε η ιστορική αλλαγή και αν, χωρίς αμετάκλητη αλλαγή των αραβικών χωρών οδήγησε στις ε, ε, ευάλωτες αυτές ε, περιόδους στην την Ισία και την Αίγυπτο και την αρχή της ευθύνης της προστασίας των πολιτών στη Λιβύα. Συνεχίζονται όμως στη Συρία, το Μπαχρέιν οι διαδηλώσεις και πρέπει να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μάθει από τα προηγούμενα στην Ισία, Αίγυπτο και Λιβύη και να μάθει ότι πρέπει να υπομίζεται τις ευθύνες της διεθνώς και εξάλλου η ευρωπαϊκή πολιτική και αυτή πρέπει να πάρει μέτρα και ε, σαρκά και Και να λάβουμε υπόψη επίση ε, τι όμορε χώρε, ώστε οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμιά ρογμή στη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ τη ελευθερία, τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχέ τη Συρία, ε, τη Ιεμένη και του Μπαχρέιν να υπενθυμηθεί σε αυτέ ότι η χρήση τη βία ει βάρο των πληθυσμών του θα έχει άμεσε επιπτώσει. Και να γνωρίζουν οι αρχέ αυτών των χωρών ότι δεν αρκούν οι εξοραϊστικές αλλαγές στα αυταρχικά καθεστώτα αυτά, αλλά πρέπει να αρχίσουν άμεσα διάλογο, ένα, μια διαδικασία διαλόγου με την αντιπολίτευση, με τα κινήματα της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας ε, των πολιτών. Πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι δημοσιογράφοι, οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να σταματήσει το, κράτος, ε, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Ευχαριστώ κυρία Μουνίθ. Περνάμε τώρα στον γύρο των παρεμβάσεων Catch the Ξέρετε ότι έχετε ένα λεπτό όλοι. Θα αφαιρέσω το μικρόφωνο αν ξεπεράσετε το χρόνο. Πρώτα, η κυρία Αντρικένε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε στην ξεκάθαρη αυτή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις τρεις αυτές χώρες. Η κατάσταση στην Συρία είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρή και ε, τα δικηβεύματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι διαδηλωτές αντικαθεστωτικοί οι οποίοι αποτελούν θύμα επιθέσεων, φυλακίσεων, συλλήψεων. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν απελαθεί από τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία ανεξαρτησία για τον τύπο. Επομένως, θα πρέπει να προβλέψουμε κυρώσεις κατά της Συρίας. Ανάλογα μέτρα θα πρέπει να λάβουμε και στην Ιεμένη και στον Μπαχρέιν. Ειδικότερα για την Ιεμένη υπάρχει μια συμφωνία για την εξαγωγή όπλων. Πιστεύω ότι πρέπει να ανασταλεί αυτή η συμφωνία. Όσον αφορά λοιπόν τι τρει αυτέ χώρε, θα πρέπει να ζητήσουμε ένα μεγαλύτερο βαθμό λογοδοσία. Δεύτερον, μια ειδική διάσκεψη τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πρέπει να λάβει χώρα. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ κύριε Άντρικεν. Τώρα ο κύριο Ροσάριο Κροσέτα, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρο. Εγώ έζησα τρία χρόνια στο Μπαχρέιν, από το 87 στο 90. Τότε το Μπαχρέιν θεωρούνταν ε, ε, μία από τις πιο δημοκρατικές χώρες του κόλπου και ακόμα συνεχίζει να ισχύει αυτό. Ε, φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία ε, κάνει δεν ξέρω πόσες ε, εκτελέσεις το χρόνο, ότι γίνονται μαζικές σφαγές, και σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχει ε, πλήρης ελευθερία του τύπου. Κάναμε αυτό το ψήφισμα για την Συρία, τον Μπαχρέιν και την Ιεμένη. Πότε θα ετοιμάσουμε όμως ένα ψήφισμα για την Σαουδική Αραβία, ε, για την Κίνα, για την ε, Αλγερία και όλες τις άλλες χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ στη Δύση είναι κάτι το περίεργο, διακόπτει ο Πρόεδρος. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Ντεσαρνέ, παρακαλώ. Ότι είναι μικρόφωνο. Δεν έχετε μικρόφωνο κύριε Κονσέτα. Η κυρία Ντεσαρνέ τώρα παρακαλώ. Ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλο τη Ευρώπη στι τρει αυτέ χώρε όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαδηλωτέ και ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα αίτημά του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε την εξή πρώτη απάντηση πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλη τη την πίεση, να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, προκειμένου να σταματήσει η καταστολή των διαδηλωτών, να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα εξολογήσει την κατάσταση και θα πρέπει να λάβει χώρα μια ειδική διάσκεψη τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τι σχέσει με τι χώρε αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ξεκάθαρα να ταχθεί υπέρ τη κοινή γνώμη, υπέρ του λαού και κατά του υφιστάμενου καθεστώτο. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα συνεχή διάλογο με όλου του εκπροσώπου τη Κοινωνία των πολιτών προκειμένου να ενδυναμωθεί η δημοκρατία, Πρέπει να προχωρήσουμε, διακόπτει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ντεσανέ. Τώρα, στη συνέχεια, η κυρία Χάουταλα, παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούσαμε ότι το Κοινοβούλιο ε, αυτή τη στιγμή το εννοεί πάρα πολύ σοβαρά ε, και θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις τρεις χώρες, τη Συρία, το Παχρέν και την Εμένη. Και πρέπει να ακούσουμε ε, τι έχουν να μας πούνε οι Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων ε, για το πώς δεν θα εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο ε, σταθμά ε, και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη ε, στο να ζητήσει ένα ειδικό μηχανισμό ε, βοήθειας προς την Συρία, τον Παχρέν και την Ιεμένη. Ε, ακούσαμε ότι είναι καιρός πια να σταματήσουμε να εξάγουμε όπλα προς τις χώρες αυτές. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, η, τι λέει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουταζα. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στην ε, Συρία οι δυνάμεις ασφαλείας ε, προχώρησαν σε χρησιμοποίηση βίας προκειμένου να καταστήλουν τους ε, διαδηλωτές. Επίσης βλέπουμε ποια είναι η στάση που υπάρχει απέναντι στο Ισραήλ, καθώς επίσης και υποστήριξη διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων. Στο Μπαχρέιν όμως βλέπουμε ότι εκεί πέρα έχουμε μια πιο μετριοπαθή μοναρχία, από την άλλη όμως έχουμε πολλούς Σιήτες, μια Σιητική αντιπολίτευση η οποία έχει την υποστήριξη του Ιράν και προχωρά ουσιαστικά σε μια προπαγάνδα κατά του βασιλιά, ο οποίος έχει προσπαθήσει να ακούσει τους διαδηλωτέ και να ξεκινήσει ένα διάλογο μαζί τους. Σαφώς βέβαια θα πρέπει να καταδικάσουμε το θάνατο όλων των αμάχων. Από ό,τι φαίνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος Σαλέχ χρησιμοποίησε βία κατά των διαδηλωτών μολονότι βέβαια έχει προσπαθήσει όλη τη τελευταία χρόνια να ταχθεί κατά της Αλκάιντα. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνο. Ο κύριος Μπρόντς παρακαλώ στη συνέχεια. Um, Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ελαφρύνουμε τα βάσανα των λαών αυτών. Τρεις προϋποθέσεις υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, ικανότητα να κάνουμε οτιδήποτε. Δεύτερον, ποιο είναι ο σωστό τρόπο να κάνουμε το οτιδήποτε. Και τρίτον, η παρούσα κατάσταση κατά κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ε, εξωτερική επέμβαση. Ε, έχουν αποδοθεί τα προβλήματα αυτά σε διεφθαρμένες κυβερνήσεις τα κράτη ε, συνήθως στέλνουν τους στρατούς τους στη μάχη να διακινδυνεύσουν ε, τη ζωή τους ε, μόνο όταν υπάρχουν ε, και διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα του κράτους αυτού. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ζωτικά συμφέροντα. Επίσης, οι εξωτερικές σχέσεις οι εξωτερικές δυνάμεις έχουν, υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον να αποσταθεροποιήσουν... Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Παουλ Ρούμπιχ παρακαλώ έχει τον λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω σε αυτές τις χώρες ζουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που νοσταλγούν την δημοκρατία, τον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία. Και αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε σε αυτές τις χώρες να κερδίσουμε φίλους και όχι συλλήβδιν να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα για αυτές. Εξατομικευμένα διαφοροποιημένα να ξεχωρίζουμε εκείνους που δεν τηρούν τους κανόνες μιας σύγχρονης κοινωνίας. Και γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να διοργανώσουμε προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δασκάλους, ε, καθηγητές, ε, δημοσιογράφους. Δουλειά μας είναι σε αυτές τις χώρες να ψάξουμε να βρούμε φίλους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ελπίζω ότι οι δράσεις με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Ολοκληρώσαμε τον παρεμβάσεων σε αυτή την περίοδο με τη κυρίας Ντότ την παρέμβαση. Παρακαλώ. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως ε, και άλλοι προαλήσαντες και εγώ συμφωνώ με μετά όσα υπόθηκαν για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την τραγική αυτή κατάσταση την οποία είδαμε σε όλη την περιφέρεια. Ωστόσο, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία που μου δίδεται προκειμένου να πω ιδίω σε εσά, κύριε Υπουργέ, ότι η δήλωσή σα σήμερα εξ ονόματο τη ύπατη εκπροσώπου για τι εξωτερικέ υποθέσει καταδεικνύει πολύ καλά, πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να πει κανεί, ότι πραγματικά είναι ανοησία το καθεστώ αυτό, η θέση αυτή και τα εκατομμύρια ευρώ που δίδονται για την θέση αυτή. Μιλήσαμε για την πρόθεση του διαλόγου, για τη μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, αλλά νομίζω ότι δεν αρκούν όλα αυτά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από ένα απλό τηλεφώνημα και από μια απλή δήλωση που ζητάει το ένα ή το άλλο. Πιστεύω ότι οι πολίτες στη Μέση Ανατολή σας ευχαριστούμε και εσάς κυρία Ντότς και ολοκληρώθηκε αυτός ο γύρος παρεμβάσεων. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο Υπουργός Νέμετ για να απαντήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου σε όλες τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Νέμετ έχει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρεμβάσεις. Καταρχήν, θα ήθελα, αν επιτρέπετε, να απαντήσω συγκεκριμένα, εξειδικευμένα σε κάποιες παρεμβάσεις για τον Μπαχρέιν. η επέμβαση του Ιράν στον Μπαχρέιν στις εσωτερικές υποθέσεις αυτής της χώρας του Μπαχρέιν αναφέρθηκε προηγούμενα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χειροπιαστά τεκμήρια μέχρι σήμερα ότι αναμίχθηκε το Ιράν στην κατάσταση στην Μπαχρέιν και ότι οδηγήθηκε η κατάσταση σε μια ριζοσπαστικοποίηση μετά από έκκληση και παρέμβαση του Ιράν. Φυσικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προβούν σε εθνικό διάλογο ε, στον Μπαχρέν οι αρχές με τους πολίτες ώστε να αποφευθεί αυτή η εναλλακτική προοπτική. Τώρα για την κατάσταση των ε, στρατιωτικών δυνάμεων και της ε, Σαουδικής Αραβίας στο Μπαχρέν. Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα έξι κράτη του κόλπου έχουν μια κοινή συμφωνία για θέματα ασφάλειας που έχουν συνάψει. Οι, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και άλλοι ζητήθηκε μέσα από το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας να παρέμβουν και να συνεισφέρουν. Και πάνω από ένα κράτος του κόλπου συνεισέφερε και ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα. Δεν είναι θέματα, ας το πω έτσι, λεπτών ε, νομικών ενιών και ξεχωριστών θα έλεγα σκιαγραφήσεων αλλά θα πρέπει να λυθούν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη οι εξελίξεις εκεί και υπό αυτό το πρίσμα να αντιμετωπιστούν. Τώρα για την Ιεμένη. Για το θέμα αυτό θα ήθελα αν επιτρέπετε να αναφέρω και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, σταματήσει να χορηγεί συγκεκριμένου είδους ε, αρρωγή προς την Ιεμένη. Για παράδειγμα, όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και σε σχέση με αυτό επιτρέψτε μου να συνεχίσω με τη μητρική μου γλώσσα για να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Σαλαφράγκα. Ο κύριος Σαλαφράγκα έθεσε το ερώτημα τι είναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της μεταβατικής περίοδου. Σε σχέση με αυτό θέλω να πω ότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση αυτής της αραβικής άνοιξης εντός εισαγωγικών. Κανείς δεν έχει την απάντηση γι' αυτό. Πριν από, πριν από κάποιους μήνες δεν γνωρίζαμε καν ότι θα υπήρχε αυτή η συνέπεια του ντόμινο που η μία αραβική χώρα μετά από την άλλη θα ακολουθούσαν αυτή την πορεία. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την αραβική άνοιξη. Γι' αυτό πολλά εξαρτώνται και από εμάς. Πολλά εξαρτώνται από τη δική μας στάση και από τις δικές μας δράσεις. Πώς αυτή η αραβική άνοιξη θα μπορέσει να έχει μια θετική έκβαση. Αυτή είναι η απάντησή μου προς τον κύριο Σαλαφράγκα. Οι προτάσεις που εξετέθησαν νομίζω ήταν πραγματικά αξιόλογες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου και της εξωτερικής διπλωματικής υπηρεσίας ή εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας όλοι τους χαιρετίζουν αυτές τις ε, ε, όλοι μας χαιρετίζουμε αυτές τις προτάσεις και όσον αφορά την πολιτική γειτονίας η εξέταση αυτής της ε, εξέλιξης αυτής της πολιτικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη Εξετάζουμε τις προτάσεις λοιπόν για αυτή την πολιτική γειτονίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια ευτυχή συγκυρία θα έλεγα σε σχέση με όλα αυτά. Γιατί αν, δεν καταφέρουμε μέσα σε κάποιες λίγες εβδομάδες σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική ε, Γειτονία να προχωρήσουμε Έχουμε δηλαδή με άλλα λόγια τον χρόνο να εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις ε, που διατυπώθηκαν για την πολιτική, ανατολική πολιτική γειτονία και να πάρουν αυτές οι προτάσεις σάρκα και ωστά. Πρέπει να είναι ενιαία, ε, να είναι εναρμονισμένη σε ένα κοινό πλαίσιο αυτή η πολιτική. Πρέπει να υπάρχει και η συνιστόσα των νότιων χωρών και όχι μόνο των ανατολικών και ιδιαίτερα πρέπει να προβληματιστούμε σε σχέση με τους νότιους ε, γείτονες μας, γείτονες των νοτιών χωρών να δούμε επακριβώς αν μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να υπάρξει μια συνετή, συνεκτική ε, πολιτική μέσα σε εναρμονισμένα πλαίσια για αυτές τις χώρες. Οι προτάσεις που διατυπώνονται σε σχέση με αυτή την πολιτική γειτονίας και ξεκινώ από το τέλος ε, και προχωρώ και μάλιστα με την κυρία Ντότς τελευταία που παρενέβη και τον κύριο Ρούμπιχε. όσον αφορά την ε, δράση για την ε, πολιτική γειτονία ε, και όλα τα συναφή στοιχεία για τη στρατηγική μας. Έχω υπόψη και τις σχέσεις με τους νέους και με την κοινωνία των πολιτών. Πραγματικά χρειαζόμαστε νέες πηγές από τις οποίες θα αντλήσουμε και στις οποίες θα βασιστούμε σε σχέση με τα διαφορετικά μεγέθη θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη ανάλογα με τη σημασία τους και ανάλογα να εμπλακούν αυτές οι συνιστώσεις. Ταυτόχρονα όμως να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο σχέσεων όπου διαφορετικές πτυχές πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι Κυρώσεις ε, εισήχθησαν, ε, θεσπίστηκαν. Απαγόρευση ε, εξαγωγής όπλων ή ανάγκη στρατιωτικής επέμβασης. Αυτό δεν μπορούσε να αποφευθεί. Και δεν κάνω λόγο μόνο για την Λιβύη εδώ, διότι δεν έχουμε μόνο την περίπτωση της Λιβύης που μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας προς τις χώρες του Νότου υπάρχει αυτή η συνιστόσα, αλλά και για την ακτή του ελεφαντοστού. Ξέρω ότι και αυτό το θέμα θα εξεταστεί, όμως αυτές τις καταστάσεις και αυτές τις χώρες δεν επιτρέπεται κανείς να συλλήβδιν ισοπεδωτικά να τις αντιμετωπίζει για τον εμφύλιο πόλεμο στην ακτή του Ελεφαντοστού ήταν κάτι το απαραίτητο να παρέμβουμε εμείς. Για αυτές τις ε, τρεις χώρες που κάνουμε λόγο τώρα εδώ, ε, για τη Συρία, την Ιεμένη, ε, τον Μπαχρέν υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα σε αυτές τις χώρες που παίζουν με την φωτιά παίζουν με τη φωτιά και υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει παρέμβαση και εκεί σε αυτές τις χώρες. Έχουμε ένα ε, πολύ σημαντικό, συγκεκριμένο και αξιόπιστο μήνυμα το οποίο απεστάλλει, το έκανε αυτό, το απέστειλε αυτό το μήνυμα, είπα τι εκπρόσωπος και είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς αυτές τις χώρες να γνωρίζουν ότι και στη Λιβύα και στην ε, ε, ακτή του Ελεφαντοστού αλλά και αλλού ότι αν χρειαστεί μπορούμε πάντα να παρέμβουμε στρατιωτικά. Στις προηγούμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα πολύ συγκεκριμένα, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο διατύπωσαν τις, ε, την αρχή της ευθύνης responsibility to protect της ευθύνης να, προστατεύσουν, να προστατευτούν οι πληθυσμοί και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να είναι κόδωνας κινδύνου που κρούεται εδώ και που πρέπει να αφουγκραστούν αυτό το μήνυμα οι, ε, οι, έχοντας, οι έχοντες την εξουσία στην ε, ε, Συρία, η Εμένη, Μπαχρέν και αλλού όπου υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα. Αυτή λοιπόν η προοπτική της στρατιωτικής επέμβασης <clears throat> δεν τίθεται σε αναλογία με το Ιράν ή το Ιράκ. Αλλά πολύ περισσότερο θα πρέπει να σκεφτούμε την περίπτωση αφρικανικών χωρών, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη και να μην το αγνοήσουν ε, οι αποδέκτες τους, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται από την Διεθνή Κοινότητα των Εθνών. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα μόνο σύντομα, α το πω έτσι υπό αναφορά κάποιων κυριότερων ενιών να παρέμβω και θα δώσω τον λόγο μετά ώστε να υπάρξει δυνατότητα να αναφερθούν οι προτάσεις σε σχέση με την είπα το εκπρόσωπο στη συνέχεια και μάλιστα σε σχέση με την σύγκληση του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Νομίζω επανειλημμένα αναφέρθηκε αυτή η πτυχή στη συζήτηση. Στην είπατε εκπρόσωπο λοιπόν θα διαβιβάσω πόσο σημαντικό το θεωρούμε το θέμα του εμπάργου όπλων να μπορέσει να εξεταστεί και να εμβαθύνουμε σε αυτό διότι θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να εξισορροπήσουμε τα πράγματα μεταξύ συνεργασίας αλλά και μεταξύ επιβολής κυρώσεων σε σχέση κυρίως με αυτές τις τρεις χώρες που ήταν αντικείμενο της συζήτησης ε, σήμερα το απόγευμα εδώ και αυτό είναι ξεχωριστή ξεχωριστός στόχος ε, αν δεν επιλέξουμε τις κυρώσεις ή τη στρατιωτική επέμβαση και επιλεγεί η ε, συνεργασία και υπάρξει η δυνατότητα να αναφερθούν κάποιες κυρώσεις σε σχέση με κάποιες χώρες αν αυτό χρειαστεί στη συνέχεια είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε η κυρία Όμεν Ρόιτεν αυτό που ανέφερε η κυρία Όμεν Ρόιτεν σε σχέση με την Τουρκία διότι και εδώ και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να τοποθετηθούμε σε σχέση με την εξέταση της πολιτικής μας όσον αφορά το μέλλον, την, το άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ελήφθησαν έξι προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έδωσαν μήνυμα ότι